Καλησπέρα. Καταρχήν, από το εξή, ο συνάδελφο Άκη Τράουστρα ε, προσεχώρησε ο κύριος Άουκε Τσούλτστρα στην ομάδα ε, ΕΝΕΦ, στην καινούργια ομάδα. Επίσης, ε, ο πρόεδρος στις 9 Σεπτεμβρίου του 2015 αποφάσισε τον κύριο Γκέρολφ Άνιμανς να τον